Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αν όχι, τι θα γίνει. Εάν είναι, κυρία Επίτροπε, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε το συντομότερο δυνατόν. Εξ ονόματος των ε, Πρασίνων Σαρτζεντίνη, η κυρία Σαρτζεντίνη για δυόμιση λεπτά.